Και θα ήθελα στην αρχή να κάνω ορισμένε παρατηρήσει αγαπητοί συνάδελφοι. Με θλίψη, καταρχήν, θα πρέπει να σα ενημερώσω ότι στο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έλαβε χώρα κοντά στι Βρυξέλλε, έχασε τη ζωή τη και η κυρία Κλάουδια Καντε, Καντεάγκο, συνάδελφο από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνία. Η κυρία Καντεάγκο εργαζόταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το Δεκέμβριο του 2008 θα διαβιβάσω εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα συλληπιτήρια και τη συμπαράσταση προς την οικογένειά της. Μια άλλη τραγωδία των περασμένων ημερών ήταν οι πλημμύρες στο πορτογαλικό νησί της Μαδέρας. Η χειρότερη θεομηνία από το 1993 που κόσε τη ζωή τουλάχιστον σε 38 άτομα. Σε αυτές τις θλιβερές λοιπόν ημέρες βρισκόμαστε με τις σκέψεις και τις προσευχές μας στον πλευρό των οικογενειών των θυμάτων των δύο αυτοκαταστροφών. Θα ήθελα τώρα να σηκωθούμε και να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των δύο τραγωδιών. Dziękuję Państwu. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να καλωσορίσω εγκάρδια τους παρόντες στην αίθουσα της Ολομέλειας, τους καλεσμένους μας από τη Λευκορωσία, την κυρία Αγγέλικα Βόρης, πρόεδρο του Συλλόγου Πολωνών της Λευκορωσίας, καθώς και τον κύριο Αλέξανδρο Μιλινκέβιτς, ηγέτη της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης και βραβευθέντα με το βραβείο Ζαχάροφ το 2006. Ο κύριος Μιλινκέβιτς είναι ηγέτης της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης στην Λευκορωσία και έχει βραβευθεί με το δικό μας